λήψης λόγου για ένα λεπτό ο κύριος Παπαστάμκος. Επιτρέψτε μου να ενημερώσω το Σώμα για την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας κατά της Ελλάδος. Οι συνεχείς παραβάσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Οι χαμηλές υπερπτήσεις μαχητικών αεροπλάνων πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά. Η παρεμπόδιση της ασφαλούς ναυσιπλοείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα και οι οχλήσεις στην έρευνα και διάσωση στην ίδια θαλάσσια περιοχή του αιγαίου που αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της ελλάδος αλλά και η εκτεταμένη προώθηση λαθρομεταναστών εκ μέρους της τουρκίας αποτελούν δυσίωνα στοιχεία για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. οφείλουμε να καταδικάσουμε την προκλητική συμπεριφορά και την συνεχιζόμενη στρατηγική αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων χώρας μέλους της Ένωσης της Ελλάδος εκ μέρους της Τουρκίας και να στείλουμε το σαφές μήνυμα ότι η συμπεριφορά της την απομακρύνει από την ευρωπαϊκή προοπτική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Τσαβαζή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για τα διακριτικά μέτρα που εισήχθησαν το 2004 που επηρέασαν τα μέλη του προσωπικού που εργάζονται ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και που προερχόταν από τα νέα κράτη-μέλη, μέτρα τα οποία θεωρήθηκαν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι ήταν παράνομο το 2008. Μετά από όλα αυτά, θέλω να τονίσω και, άλλο, και άλλη διακριτική απόφαση που είχε αποτέλεσμα διάκριση. 4,5 χρόνια μετά βρίσκουμε ότι αυτοί οι πολίτες των νέων κρατών μελών ακόμα θεωρούνται σαν πολίτες ε, δεύτερης κατηγορίας, από κράτη-μέλη δεύτερης κατηγορίας. Τι συνέβη κύριε Πρόεδρε, πέρσι διαφημίστηκε, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για επικεφαλή μονάδας που θα ήταν υπεύθυνο για τους Ούγγρους διερμηνείς που εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολίτες από κάθε Ευρω... κράτος Ευρωπαϊκής Ενώσεως είχαν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Ο επικεφαλής της μονάδας έχει συντονιστικά ε, καθήκοντα και πέραν αυτού επικεφαλής της μονάδας επίσης παίζει σημαντικό ρόλο εξασφαλίζοντας το ότι η ειδική ορολογία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αντικατοπτρίζεται σωστά στην ουγγρική γλώσσα. Είχαμε δύο ψηφίους, ε, έναν με μητρική τα αγγλικά και έναν με μητρική τα ουγγρικά. Και εκπλήσωμε διότι βλέπω ότι τελικά ο υποψήφιο με μητρική τα αγγλικά προτιμήθηκε. Φαντάζεστε αν ο Γάλλος επικεφαλής μονάδας να ήταν Ισπανός να έχει αμυντική δεσπανικά. Αυτή είναι διακριτική μεταχείριση, είναι απαράδεκτη και θα δημιουργήσει σοβαρέ ζημιέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα έγγραφα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, τη μετάφραση των εγγράφων στι διάφορε γλώσσε. Και εκ μέρου όλων των νέων κρατών μελών θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ κατά αυτή τη αποφάσεω. σα ευχαριστώ πολύ. Θα λάβετε ασφαλώ απάντηση. Ακολουθεί ο κύριος Κρίστιαν Σίλβιου Μπουζόη. Christian It's Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα το απόγευμα ακούσαμε εσά και άλλου. Κάνατε δηλώσει για τη φρικτή κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη που υπάρχει για άμεση κατάπαυση του πυρός και την απόσυση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τη Γάζα. Πρέπει να πω ότι σε αυτό το πλαίσιο συμφωνώ με τον κύριο Γκον ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τοποθετηθεί. Δεν μπορούμε να μην ήμασταν αποφάσιστοι. Αλλά τώρα τι να μιλάμε για καθημερινά θέματα όταν έχουμε ακούσει όλα αυτά. Αλλά βέβαια καθημερινά θέματα αφορούν όλου του πολίτε. Και στην Ιρλανδία ανακοινώθηκε από την ΤΕΛ ότι 2.000 θέσει εργασία θα μετακινηθούν. Και αυτό έπληξε την κοινότητα στην Δυτική Ιρλανδία. Όταν έχουμε κρίση, αυτό δημιουργεί ιδιαίτερε δυσκολίε στου εργαζομένου που απασχολούνται από την ΤΕΛ και για εκείνου που παρέχουν διάφορα υλικά στην ΤΕΛ. Σε αυτό το πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίηση θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να βοηθήσει την επανακατάρτιση των εργαζομένων και θα πρέπει να προωθηθεί και το πνεύμα του επιχειρήν για την αυτοαπασχόληση. Θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση αμέσω να υποβάλει αίτηση στο Ταμείο Παγκοσμιοποίηση, ώστε εργαζόμενοι να έχουν κάποια εμπιστοσύνη στο μέλλον και να δουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται τόσο ώστε να βοηθήσει όσου εργαζομένου σε αυτή την περίπτωση εκείνου που είναι στα, Μεσοδυτική Ιρλανδία και τη Δυτική Ιρλανδία. Ακολουθεί Ρίτσαρτ Τσαρνέτσκι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Μετά από τη σύναψη μιας ε, συμφωνίας, συμφωνίας για την αποστολή του ρωσικού φυσικού αερίου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, φαίνεται ότι συνήφθη συμφωνία, αλλά πού είναι το φυσικό αέριο. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταδείξουν αλληλεγγύη κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ε, παρόλα αυτά όμως, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το μόνο που λείπει είναι η αλληλεγγύη από αυτή τη διαφωνία, διότι πολλά κράτη-μέλη ακολούθησαν διαφορετική θέση και στο τέλος αποφασίσαμε να ευθυγραμμιστούμε κάπως, να ακολουθήσουμε μια κοινή θέση. Ξέρω ότι θα το συζητήσουμε σε δύο μέρες, αλλά θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί ένα οικονομικό μέσο για πολιτικούς σκοπούς και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια κοινή ενεργειακή πολιτική και όχι μια ενεργειακή πολιτική που να ορίζουν τα μεγάλα κράτη-μέλη που χτίζουν φυσικούς αγούς κάτω από τη Βαλτική. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωρίζουμε ότι η Coca-Cola και τα πατατάκια είναι κακά για την υγεία μας. Και στο παγκοσμιοποιημένο μας περιβάλλον γνωρίζουμε ότι και άλλα προϊόντα είναι προβληματικά αλλά έγιναν διάφορες δηλώσει για το κρασί Φερρυπίν και στην περιοχή μας παράγουμε κρασί. Δίδονται χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως σε εκείνου που αποφασίζουν να μην συμμετέχουν πλέον στην παραγωγή κρασιού. Στην κοιλάδα των Καρπαθίων έχουμε ιστορική παράδοση. Στην Ουγγαρία είχαμε πολύ καλή παραγωγή ίνου. 600.000 εκτάρια καλλιεργούνται για την παραγωγή ίνου. Το 1948, ακόμα και τότε, παράγαμε κρασί στα 200.000 εκτάρια. Σήμερα 40.000 εκτάρια καλλιεργούνται αμπέλια για κρασί. Λοιπόν, για την περιοχή των Καρπαθίων θα πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται. Καταστράφηκε η παραγωγή του κρασιού σε αυτή την περιοχή. Οι Ούγγροι πιστεύουν στην καλή υγεία και στο καλό κρασί και σας εύχομαι καλή χρονιά λέγοντας αυτά. Κύριε Μακδόναλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για την Παλαιστίνη θέλω να μιλήσω. Κύριε Πρόεδρε, στα σχόλιά σας προηγουμένως, ε, ήσασταν προσεκτικό στην τοποθέτησή σας έναντι του Ισραήλ. 900 Παλαιστίνοι είναι νεκροί. Ένα τρίτο από αυτούς τους νεκρούς είναι παιδιά. Και δεν μπορούμε να βρούμε το κουράγιο σε αυτή την αίθουσα να το κουράγιο να, καταδικάσουμε την ομότητα του Ισραήλ. Και αυτή η επίθεση δεν είναι μόνο δυσανάλογη, είναι και εντελώς αδικαιολόγητη. Δεν είναι οι ανάγκες του Ισραήλ που οδηγούν σε αυτή την απόφαση. Είναι κοινική, κλινική επίθεση, όχι κατά της Αμάς, αλλά κατά του Παλαιστινιακού πληθυσμού. Και νομίζω ότι τα κράτη-μέλη έχουν ηθική υποχρέωση να ασκήσουν διπλωματική και πολιτική πίεση εναντί του Ισραήλ για να λήξει αυτή η βία. Τώρα να χαϊδεύουμε την Ισραηλινή κυβέρνηση είναι κάτι που δεν θα δουλέψει. Ποτέ δεν δούλεψε αυτό. Και το Ισραήλ πρέπει να καταλάβει τώρα ότι υπάρχουν συνέπειες για τις δράσεις του. Καλό όλους τους ευρωβουλευτές λοιπόν να απαιτήσουν την άμεση ε, αναστολή της συμφωνίας της Ευρωμεσογειακής και όλων των προτιμησιακών εμπορικών διευθετήσεων και συμφωνιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ. Εξίσου θα πρέπει να αντισταθούμε κατά ιασδήποτε απόπειρα να αναβαθμιστούν στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του κράτους του Ισραήλ που πολιορκεί την Γάζα και βιοπραγεί κατά των Παλαιστινίων. Η όλη ρητορική για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ακούγεται συχνά σε αυτή την αίθουσα θα πρέπει να μεταφραστεί πράγματι σε πράξεις αυτή είναι η μόνη προοπτική, κύριε Πρόεδρε, για επιτυχή ρηνευτική διαδικασία στην Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστώ. Και από τον χρόνο και μόνο που ε, χρησιμοποιήσατε, που ήταν το διπλάσιο ε, του λεπτού, ε, φαίνεται πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα αυτά και πόσο δύσκολα πάντα συμπτύξει κανεί ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάντω για την παρέμβασή σα. Η εκλογική μου περιφέρεια, ξέρετε, έχει πληγεί διότι χάθηκαν 2.000 θέσεις εργασίας σε εργοστάσιο και αυτό σημαίνει ότι θα χαθούν και άλλες 2.000 που εξαρτώνται από την ΔΕΛ. Η ΔΕΛ θα κινηθεί στο Λόντς στην ε, Πολωνία και δόθησαν 52 εκατομμύρια ως ε, κρατική επιδότηση. Αυτά εντάσσονται στους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα δοθούν κονδύλια για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης και αυτού του φαινομένου όπου χάνονται θέσεις εργασίας σε ορισμένα γεωγραφικά σημεία. Ακολουθεί ο κ. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Δύο μέρες πριν τέσσερα σχολεία στο Μπουργκάς αντιμετώπισαν συνθήματα που είχαν ε, συνθήματα στους τοίχους που μιλούσαν για θάνατο στους γκάουερς. Αυτό χρησιμοποιόταν κατά την ε, τουρκική, την οθωμανική, τους οθωμανικούς καιρούς, που, όπου αυτή η κατηγορία ε, θεωρείται σαν να επρόκειτο για υπανθρώπους. Η ίδια λέξη gowers, χρησιμοποιήθηκε από, και από τον πρώην Υπουργό Γεωργίας. Θα ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την ε, ορολογία. Όπως ξέρετε, η Τουρκία δεν έχει καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι είναι κατά της ισότητας. Υπάρχει δυστυχώς μισαλοδοξία εθνοτική μισαλοδοξία Εμείς ήμασταν κατά αυτών των τάσεων και νομίζω ότι θα πρέπει να, να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαίρω τη Τσεχική Προεδρία της προσπάθειας που κάνει να αντιμετωπίσει την κρίση με το φυσικό αέριο. Αλλά διαμεσολάβηση σε διαδοχικές κρίσεις δεν είναι λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμείνει σε ρόλο γκουβερνάντας ενός άταχτου παιδιού. Ποιο είναι το σαφές συμπέρασμα. Χρειάζεται στρατηγική συμμαχία με τη Ρωσία που θα παρέχει ενέργεια. Αλλά αυτή η προσέγγιση τελικά είναι λανθασμένη η αιτία τη κρίσεω δεν είναι η Ουκρανία, αλλά είναι εντός των κόλπων της Γκάσπρομ, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσει τη. Διότι για 8 διαδικτυακά χρόνια η παραγωγή φυσικού αερίου της Γκάσπρομ είχε αποτελεματωθεί στα ίδια επίπεδα. Τυπικό αποτέλεσμα πολιτικού κρατικού ελέγχου στην παραγωγή. Δεν μπορεί να δώσει αέριο και στους Ρώσους και στο εξωτερικό. Και έτσι ο κ. Ε, δημιούργησε αυτή την πολιτική κρίση. Και τελικά αποδιοπομπαίος τράγος είναι η Ουκρανία. Άρα πολύ πιο σημαντικό τώρα εμείς να επικεντρώσουμε στις προσπάθειές μας επί της εξευρέσεως νέων πηγών ενεργείας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Als nächste Magda Kosane Kovac. Kosane Kovacs. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε, που ε, θεωρούσαμε ότι είχε καθαρά ε, λόγους ε, δημαγωγικούς, δημαγωγικής προβολής, βλέπουμε ότι πλήττει τους πάντες, τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματίες, όλες τις κοινωνικές τάξεις. Είχαμε μία ανακοίνωση της Επιτροπής επί του θέματος και βλέπουμε ότι δεν βρισκόμαστε όλοι στην ίδια κατάσταση. Υπάρχουν αυτοί που βρίσκονται στα περιθώρια της κοινωνίας, στα περιθώρια της Ευρώπης και έχουν πληγεί ακόμα περισσότερο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την αξιοποίηση εργασία και επίσης δεν θα πρέπει να έχουμε αναζωπήρωση της φτώχειας στην Ήπειρό μας. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε πόρους, γι' αυτό και θα ήθελα να καλωσορίσω την της Επιτροπής και του Επιτρόπου Σπίτλα, ο οποίος τόνισε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις πιο ευάλωτες κατηγορίες για να τις υποστηρίξουμε σε αυτή την ε, περίοδο φθήνουσας οικονομικής πορείας. Ελπίζω να έχουμε μια αντίδραση από πλευράς της Επιτροπής έτσι ώστε να μην υπάρχει εξαναγκαστική ομοιομορφία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς να συμμετάσχουμε σε αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κύριος Μάγκορ Τσίμπι. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Βλέπουμε ένα παράδοξο. Να είναι αντίθετοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές με τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, παρόλα αυτά να τα προτιμούν όταν τα βλέπουν στα σούπερ μάρκετ. Αυτό οφείλεται ωστόσο και στο ότι είναι επισημασμένα με ετικέτες τα οποίε δεν είναι βαναγνωστές. Το σωστό θα ήταν οι ετικέτες να γράφουν καθαρά, αλλά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι απαραίτητες διατάξεις και δεν υπάρχει ε, δυνατότητα, μάλλον οι χώρες μέλη έχουν τη δυνατότητα επιλογής. Ορισμένες χώρες έχουν περιλάβει σχετικές διατάξεις, άλλες δεν δέχονται να δίνεται η πληροφορία αυτή. Οι καταναλωτές ωστόσο θέλουν να μπορούν να επιλέγουν τα τρόφιμα ανάλογα με τις δικές τους αξίες. Εάν μας ενδιαφέρουν πραγματικά οι ανησυχίες των καταναλωτών, τότε πρέπει να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και να τους δώσουμε τη δυνατότητα επιλογής. Γι' αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ώστε θα μπορέσουν, να μπορέσουν όλες οι χώρες να επιβάλλουν τις σχετικές διατάξεις για την επισήμανση των τροφίμων αυτών. Ο κ. Κογκάλσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλέσω το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 13 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να λάβει μέτρα. Να λάβει μέτρα κατά διακριτικής μεταχείρισης για λόγους εθνοτικής καταγωγής. Δύο από τους τρεις Λιθουανούς πολωνικής καταγωγής που εξελέγησαν στο Λιθουανικό Κοινοβούλιο κινδυνεύουν να στερηθούν τα προνόμια τους και να χάσουν τη θέση τους με την αιτιολογία ότι είναι εθνοτικοί Πολωνοί, έχουν πολωνική καταγωγή. Είναι παράλογη και σκανδαλώδης η κατάσταση, είναι διάκριση για εθνοτικούς λόγους και δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων με έναν τρόπο που είναι απαράδεχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Vielen Dank. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, συνάδελφοι, ο Μπέντ Πόσελτ εκπροσωπεί το CSU της ε, Βαβαρίας και είναι επικεφαλής του Landmannschaft της Ουδετίας και κάλεσε την Τσεχική Προεδρία την Τσεχική Δημοκρατία να αναστείλει το διάταγμα Μπένες κατά διάρκεια της Τσεχικής Προεδρίας. Αυτές οι διακηρύξεις Μπένες υιοθετήθηκαν όμως σε μια προσωρινή ενδιάμεση περίοδο. Είναι παράδεκτο αυτό το αίτημα. Όταν δεν υπήρχε κανονική κυβέρνηση. Δεν είναι καρκίνωμα όπως αναφέρει αν κάποιο είναι καρκίνωμα, είναι εκείνο που ε, ε, έστρεψε τέτοιε επιθέσει κατά τη ε, τσεχική δημοκρατία. Δεκάδε χιλιάδων Γερμανών ζουν στην τσεχική δημοκρατία και πολύ περισσότεροι την επισκέπτονται. Και είναι πολύ ικανοποιημένοι οι Τσέχοι που ζουν στη, Γερμανία. Εγώ εξελέγην Ευρωβουλευτή παρά το γεγονό ότι είναι Ευρωπαίο πολίτη, ε, συγγνώμη, Γερμανό πολίτη, εξέλεγει στην ε, Τσεχία. Πρόεδρε, η κρίση του φυσικού αερίου άφησε εκατοντάδε χιλιάδε ε, νοικοκυριά σε 17 κράτη μέσα τη Ευρωπαϊκή Ενώση χωρί τέρμανση σε τέτοιε χαμηλέ δημοκρασίε στην Ανατολική Κεντρική Ευρώπη. Επλήγει περισσότερο από τη διαφορά αυτή, τη διένεξη που έκλεισε εργοστάσια και σχολεία. Ακόμα και αν το Κίεβο και η Μόσχα υπογράψουν τη συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από ώρε συζητήσεων με του Ευρωπαίου, η Gazprom λέει ότι για να ξαναρχίσει την παροχή αερίου μέσω Ουκρανία θα καθυστερήσει, διότι δεν έχει λάβει αντίγραφο τη συμφωνία. Μία ομάδα εμπειρογνωμών που απεστάλλει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει ποιε είναι οι ροέ από τη Ρωσία προ την Ουκρανία. Και ακόμα αν αρχίσει η ροή φυσικού αερίου στην Ουκρανία θα χρειαστούν 36 ώρε, μέχρι 36 ώρε να φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν αποτέλεσμα αυτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια νέα πολιτική όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό τη, ώστε να αποφευθούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον και θα πρέπει να υπάρχει ποικιλία ενεργειακών πηγών. Καλωσορίζω την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαφορά αυτή, στη ένεξη αυτή και ελπίζω ότι μια συμφωνία τελικά θα επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατόν, ούτω ώστε να αποφευθεί ε, μια αύξηση, μεγέθυνση τη κρίσεω. Γιούρι. Αουρέλιο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Πέρσι, όπως ξέρετε, είχαμε πανηγυρίσει τον τέταρτο χρόνο πυρηνικού αφοπλισμού. Νωρίτερα είχαμε εγκρίνει ένα ψήφισμα όπου ο πρόεδρος της Επιτροπής και το Συμβούλιο τόνισαν ότι θα προωθήσουν τις πολυμερείς συμφωνίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να, ε, μάλλον να ελέγξουμε την συνθήκη. Ξέρετε ότι δεν σταθήκαμε επιτυχής σε αυτό μας το εγχείρημα και χρειάστηκε τα Ηνωμένα Έθνη να ξαναεξετάσουν το ζήτημα αυτό. Όταν το ήλθα στο κοινοβούλιο αυτό το Νοέμβριο. Και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη, δηλαδή αυτές οι εξελίξεις και έχουμε πραγματικά σταθεί επιτυχής. Γνωρίζουμε για την πυρηνική ασπίδα στη Τσεχική Δημοκρατία και την Πολωνία και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση, αρνητική κλιμάκωση σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Νικολέσκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά ελέγχθησαν για την ε, κρίση στον τομέα του φυσικού αερίου και όλοι ανέφεραν ότι είναι πολύ επικίνδυνο το γεγονός ότι εμείς εξαρτόμαστε άμεσα από τη Ρωσία και την παροχή φυσικού αερίου. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια διαφοροποίηση και να βρούμε άλλες εναλλακτικές ε, πηγές ενέργειας. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι κατασπαταλούμε την ενέργεια γιατί το 1 τρίτο της κατανάλωσης είναι, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ε, κατασπατάλης και εμείς εισάγουμε στη Ρουμανία 14 εκατομμύρια τόνων αντίστοιχων τόνων πετρελαίου και δυστυχώς ένα εκατομμύριο κατασπαταλάτε διότι δεν υπάρχει σωστή μόνωση στα σπίτια μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν βελτιώνει αυτή την κατάσταση διότι δεν προβλέπει χρηματοδοτήσεις ιδιαίτερα στον τομέα της μόνωσης. Τι είναι ευκολότερο να βρούμε νέες πηγές ενέργειας ή θα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι με απλά μέτρα μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Als Μίλος Κότερεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, φέτος θα ασχοληθούμε με την ε, δέκατη επέτειο της χρήσης του ευρώ. Όπως ξέρετε, η Σλοβακία έγινε πλήρες μέλος την 1η ε, Ιανουαρίου. Εμείς ε, τηρήσαμε όλες τις προδιαγραφές σε σχέση με το εθνικό μας νόμισμα, αλλά τώρα έχουμε εγκρίνει το ευρώ. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργό ε, Βίτσο, το ευρώ είναι ένα νόμισμα το οποίο μπορεί να μας προστατεύσει κατά πολλών κινδύνων και να βοηθήσει την Σλοβακία να ανθίσει. Θα ήθελα να συγχαρώ τους Σλοβάκους για την θετική τους στάση έναντι του κοινού νομίσματος και τους εύχομαι κάθε επιτυχία μέσα στα πλαίσια μιας ευημερίας. Η κυρία Παναγιωτοπούλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, επειδή δεν θα γίνει σχετική συζήτηση στο Κοινοβούλιο, ε, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση η πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές. Πρόκειται για την εργασία των ναυτικών σύμφωνα με τη Σύμβαση της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Έτσι, η ναυτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας ε, και είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να δοθεί σχετική όθηση. Ε, από εκεί περιμένουμε ανάπτυξη και παραγωγικότητα. οι θάλασσες που βρέχουν την ευρωπαϊκή ένωση είναι θάλασσες που είναι σημαντικές για το διεθνές εμπόριο και ε, πιστεύουμε ότι οι νέοι πρέπει να δουν το μέλλον τους στη θάλασσα και να πλαισιώσουν την ε, ναυτιλία. Ευχαριστώ. Äh, Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, από αρχές Οκτωβρίου 2008 ζητώ να λάβω λόγο σε αυτές τις παρεμβάσεις του ενός λεπτού και ε, χαίρομαι πάρα πολύ που επιτυγχάνετε τώρα. Ενώ, για παράδειγμα, ε, έχω ακούσει τρεις φορές τον κύριο Ρογκάλσκι. Τώρα, επί της... Ε, υπήρχε, η αστυνομία στην Αυστρία σταμάτησε ένα, με παράνομο εμπόριο και μεταφορά ζώων, σκύλων στην Αυστρία όπως είπα που υπονομεύουν ή ε, καταστρατηγούν τις σχετικές διατάξεις. Χρειαζόμαστε κοινή νομοθεσία και κοινέ προδιαγραφές για όλη την Ευρώπη, οι οποίες να πρέπει και να μπορούν να επιβάλλονται από όλες τις χώρες μέλη. Γιατί μέχρι τώρα οι αρχές έχουν μείνει άπραγες. Σας ευχαριστώ. Κατσίν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, οι σφαγές, οι αιματηρές των Παλαιστινίων στη Γάζα είναι ένα σύμβολο της κακής δουλειάς που κάνουμε. Πρέπει πραγματικά να έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς Παλαιστινίους μπροστά μας πριν τα θεσμικά όργανα να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι είναι φορέας διεθνών σχέσεων και σημαντικός πολιτικός πρωταγωνιστής. Είμαστε πραγματικά. Ο Ισραηλινός στρατός επιτίθεται κατά σχολείου γεμάτου πολίτες που χρηματοδοτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σωστό αυτό. Δεν υπάρχει ανθρωπιστικό δίκαιο κατά της ε, μετακίνηση Παλαιστινίου σε ένα σπίτι και το σπίτι να βομβαρδίζεται την επόμενη μέρα. Ξέρω πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτές οι Ισραηλινέ δράσει είναι δυσανάλογες και απάνθρωπες. Οι δράσεις τους είναι ανήθικες, στρεβλέ και παράξενες. Διότι μόνο και μόνο γίνεται προεκλογική εκστρατεία. Είναι μια αιματηρή προεκλογική εκστρατεία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δράτω με τι ευκαιρίε να πω ότι πρέπει να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους ειδικού Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Βαρσοβία το 2010. Οι ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες που διεξήχθησαν στην θα διεξαχθούν στην Αθήνα το 2011. Έδωσε 5 εκατομμύρια ευρώ για τους ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στην Ιρλανδία το 2003 και ήταν υπέροχη ευκαιρία και χαρά για πάρα πολλού που ήμασταν παρόντε. Εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή υποστηρίξεω των εθελοντών για τον αθλητισμό. Κύριε Πρόεδρε, να προσθέσω ότι υπάρχει γραπτή δήλωση για αυτό το θέμα που οι ευρωβουλευτέ μπορούν να υπογράψουν αυτή την εβδομάδα εκτό τη αίθουσα Ολομέλεια και παροτείνω όλου του συναδέλφου να υπογράψουν αυτή τη διακήρυξη για την υποστήριξη ευρωπαϊκή χρηματοδοτήσεω για αυτού του πολύ σημαντικού ειδικού Ολυμπιακού Αγώνε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γιάρομιε Κόλιτσεκ. Καλή χρονιά κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη βαθιά μου έκπληξη για τον παράδοξο τρόπο με τον οποίο η τσεχική δημοκρατία που είναι γνωστή για συγκεκριμένη στάση της όσον αφορά την αντιμετώπιση της Ρωσίας απέτυχε να βρει τη σωστή προσέγγιση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ήταν μια χώρα που δεν ήθελε να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία για, την, για τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό και συγκλονίζομαι και από την στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κύριο Κομπέντιτ που απειλούν τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία με την επιβολή κυρώσεων αν αυτές οι χώρες τελικά ενεργοποιήσουν τους πυρηνικούς τους σταθμούς. Αυτό ήταν κακό αστείο ή θα πρέπει τελικά να δείξουν αυτοί οι αλληλεγγύοι, αυτοί οι άνθρωποι εκεί που παγώνουν. Ο κύριος Αγγελάκας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αναφερθώ και εγώ στο θέμα του φυσικού αερίου που τις τελευταίες δέκα μέρες γινόμαστε μάρτυρες της διαμάχης γύρω από το θέμα αυτό. Μια διαμάχη που έχει φέρει σε ομοιρία πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξαρτώνται ενεργειακά από το φυσικό αέριο και έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πολίτες, επιχειρήσεις και βιομηχανία μέσα από συζητήσει των δύο αντιμαχόμενων πλευρών που χαρακτηρίζονται από καχυποψία κακοπιστία και αλληλοσυγκρουόμενε ανακοινώσει και με την παρέμβαση της ευρωπαϊκής προεδρίας και της επιτροπής φαίνεται πως βρέθηκε κάποια λύση. είναι φανερό ότι ανεξαρτήτως προθέσεων και καταμερισμού το πρόβλημα μπορεί να ξαναπροκύψει εάν δεν ληφθούν μέτρα πρέπει λοιπόν να μελετηθεί η αναδιατύπωση του ενεργειακού δόγματος της ευρωπαϊκής ένωσης με την προσθήκη σε αυτό και άλλων πηγών ενέργειας. θα πρέπει επίσης το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με σαφήνεια να στείλει το μήνυμα ότι η ευρωπαϊκή ένωση δεν εκβιάζεται και να συμμετάσχει στη συζήτηση για το σχεδιασμό εναλλακτικών οδών για ασφαλή και συνεχή παροχή φυσικού αερίου ο στόχος της μείωσης των ενεργειακών αναγκών κατά 20% μέχρι το 2020 δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν η σημερινή κατάσταση είναι τόσο ασταθής και όχι δεδομένη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω την κυρία Λίνεμαν. Η κυρία Σίλβια Αντριάννα Τικάου δεν νομίζω... Α, είναι παρούσα η κυρία Τικάου. Έχει το λόγο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ως προτεραιότητα να θέσει μια κοινή ενεργειακή πολιτική και ένα κοινό ενεργειακό σχέδιο και πρόγραμμα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Οι περικοπές παροχής φυσικού αερίου δείχνουν ότι είμαστε άμεσα εξαρτώμενοι από ε, εξωγενείς πηγές και οι χαμηλές θερμοκρασίες φέτος δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, μία στρατηγική στα πλαίσια και του, του ενεργειακού τομέα για να φτάσουμε σε μία διαφοροποίηση πηγών. Στα πλαίσια του υγροποιημένου, ε, του, του υγροποιημένου, υγροποιημένης μορφής ε, μορφών ενέργειας, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και το σύστημα αγωγών. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με την ΕΤΕ και με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να εξευρεθεί επαρκής χρηματοδότηση. Σε το λόγο τώρα για ένα λεπτό. Uh, um, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι θέλω να θίξω το θέμα της Ζιμπάμπουε. Νομίζω ότι αν δεν δούμε κάτι στην τηλεόραση δεν ε, βλέπουμε τα προβλήματα που ανακύπτουν εκεί. Είδαμε φέτος ότι ένα μέλος ε, μιας μη κυβερνητικής μας, ε, δεν γνωρίζαμε μάλλον την τύχη του για 21 μέρες πριν βρεθεί στο Χαράρε και ίσως ε, τον κακομεταχειρίστηκαν και τον βασάνισαν επειδή τάχτηκε υπέρ των, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κυρία Μακόκο, όπως ξέρετε, βρίσκεται σε δυσχερή θέση και σε κατοίκον περιορισμό και δυστυχώς βρίσκεται στα χέρια της ε, κυβέρνησης, απάνθρωπης κυβέρνησης Μουγκάμπε. Πολλά συζητήθηκαν εδώ, μιλάμε για ένα εφιάλτη για τους κατοίκους της Ζιμπάμπουε και πιστεύω ότι θα πρέπει και εμείς να επανεκφράσουμε το ενδιαφέρον μας έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη τις εγκληματικές δραστηριότητες κατά των ανθρώπων και των ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Ντερόσα τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαιρετίζω τη δήλωση του Προέδρου που αναφέρθηκε στη Γάζα και χαιρετίζω και την απόφαση του Κοινοβουλίου για ψήφισμα επ' αυτού που θα ζητεί άμεση μόνο με κατάπαυση του πυρός που θα γίνει σεβαστή από όλες τις πλευρές στη Γάζα. Πάνω από 900 νεκρούς έχουμε. Η ματαιότης τη διαμόρφωση πολιτική μέσω του πολέμου είναι προφανέστατη. Θα πρέπει να επιμείνουμε το Ισραήλ να σταματήσει του φόνου. Η Γάζα είναι η μεγαλύτερη φυλακή στον κόσμο. 1,5 εκατομμύριο φυλακισμένου έχει και επίσης δυστυχώς είναι σφαγείο τώρα. Άντρες, γυναίκες και παιδιά πεθαίνουν απλώς διότι είναι Παλαιστίνοι. Τι πιθανά εγκλήματα έκαναν τα παιδιά των Παλαιστινίων που πεθαίνουν σε αυτή την σύγκρουση τι δικαιολογία έχουμε εμεί οι Ευρωπαίοι να εξακολουθούμε να συνάπτουμε εμπορικέ συμφωνίε με του Ισραηλινού όταν σφάζει του τους Παλαιστινίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να πάψει να προβάλλει δικαιολογίε, να πάψει να τσακώνεται και με μια ενιαία δράση να σταματήσει τη σφαγή. Δεν μπορούν να βαθμιστούν οι σχέσει τη Ευρώπη με το Ισραήλ από τη στιγμή που το Ισραήλ δεν ξεκινά επικοδομητικά διάλογο με όλου του εκπροσώπου των Παλαιστινίων. Ευχαριστώ. Ξεπεράστε λίγο το χρόνο βέβαια. Η κυρία Φόλτιν Κουμπίτσκα έχει το λόγο. Για ένα λεπτό σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός χωρών που βασίζεται σε κοινέ αξίες και θα κάνει τα πάντα για να σταματήσει η προβολή, η πρόθεση του μίσους. Η Utelsat, η γαλλική εταιρεία, αποφάσισε να εκπέμψει ε, ένα κανάλι της Χαμάς το οποίο κανάλι ε, στρέφεται κατά των Ιζαρινών. Η Eutelsat έδειξε για μία ακόμη φορά ότι οι επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν υπόψη δεοντολογικά στοιχεία ηθική. Ο αυτός, ο NDTV της, της Κίνας, έχει μπλοκαριστεί. Δεν εκπέμπει. Παρά τις διαμαρτυρίες, το Διοικητικό Συμβούλιο της UTELSAT αρνείται να αλλάξει απόφαση όσον αφορά το κινέζικο κανάλι. Το Διοικητικό Συμβούλιο της UTELSAT είναι πολύ παράξενο. Δεν ξέρω πώς παίρνει αποφάσεις. Για ένα λεπτό, μη Η κυρία Φιγκεϊρέδο. Α, όχι. Θα ήθελα να η κυρία Φιγκερέδο έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η επίθεση του Ισραήλ κατά της Γάζας αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Μιλάμε για 900 Παλαιστίνιους που έχουν ήδη πεθάνει, μεταξύ των οποίων άμαχοι και παιδιά θα πρέπει να επιμένουμε για την πάυση του πυρός και για την πάυση του αποκλεισμού αυτού. Γιατί μιλάμε για ένα απέραντο στρατόπεδο στο οποίο έχει μετατραπεί με η λωρίδα της Γάζας. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την έντονη αντίδραση όλων των κρατών, διότι όλοι μιλάνε για τον τερματισμό αυτό του τεράστιου εγκλήματος. Πιστεύω ότι όλοι οι υπεύθυνοι οργανισμοί θα πρέπει να απαιτήσουν την άμεση κατάπαυση του πυρός καθώς και την άρση του αποκλεισμού. τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σβερίνα. Σβερίνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόσφατα μου έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι οι τσεχικές ασφαλιστικές εταιρείες δεν δίνουν ένα ε, ειδικό πριμ στις γυναίκες που ζητούν την ασφάλιση στα πλαίσια δηλαδή της ασφάλισης αυτοκινήτου. Βλέπω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μία διάκριση Βλέπουμε ότι ορισμένοι πολιτικοί και μη κυβερνητικέ αντιμετωπίζουν το ζήτημα που οδηγούν ένα σκεπτικό στα άκρα του. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την αναλογιστική που μας δείχνει ότι οι γυναίκες συμπεριφέρονται διαφορετικά ως οδηγοί από τους άνδρες και θα ήταν γελίο να θεωρήσουμε ότι συμπεριφέρονται κατά τον ίδιο τρόπο. Αντιδρούν διαφορετικά και υπάρχουν βιολογικοί λόγοι ε, γι' αυτό. Έχει το λόγο. Uh, thank you, Madam President. ευχαριστώ. Μία νέα δημοσκόπηση, δημοσκόπηση έχει δημοσιευτεί στη Μεγάλη Βρετανία και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 83% θα ήθελαν ε, να υπερέχει το εθνικό μας δίκαιο και να μην δεσπόζει το κοινοτικό. Το 71% θέλουν ε, μία, να γίνει ένα δημοψήφισμα έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο θα ισχύσει η συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Οι Βρετανοί θέλουν το ελεύθερο εμπόριο, ε, φιλία και συνεργασία με την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, όχι να διέπονται απόλυτα από τις αρχές Ευρώπης. Εάν γίνει ε, μία πραγματική αν ε, λάβουμε υπόψη αυτή την τάση, τότε οι περισσότεροι θα ζητούσαν να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. το λόγο. Ε, Κυρία Πρόεδρε, να εκφράσω ανησυχίες για την αυξανόμενη έλλειψη επιστημονικών στοιχείων στα σχέδια προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που του στο Κοινοβούλιο και σε κάποιες εκθέσεις και τροπολογίες για τις οποίες είμαστε εμείς υπεύθυνοι βουλευτές. Η σωστή επιστήμη υποχωρεί σε λαϊκιστικές απαντήσεις που καλύπτονται στα πλαίσια της αρχής της προλήψεως, όπως ε, τα φυτογενομικά προϊόντα. Ε, τα αξιολόγηση κινδύνου απαγορεύεται. Δεν γίνεται αξιολόγηση κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει επιστημονικός ε, ορισμός των οσιών που επηρεάζουν ενδοκρινικές λειτουργίες και δεν υπάρχει και σωστή, σωστός προσέγγιση προσέγγισης με την οδηγία REACH η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως χάνει την αξιοπιστία της. Διότι όλο και περισσότερο η σωστή επιστημονική προσέγγιση απουσιάζει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπίνεφ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η κρίση του φυσικού αερίου που έπληξε την Ευρώπη τώρα αρχάς του 2009 έχει λάβει ε, καταστροφικές διαστάσεις για τη Βουλγαρία. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές ε, για την ε, παροχή φυσικού αερίου, την προμήθεια φυσικού αερίου στη Βουλγαρία από πηγές Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι βραχή, είναι λάθος η απόφαση των Βουλγάρων ηθινόντων να καταστήσουν τη Βουλγαρία απολύτως εξαρτημένη από την παροχή φυσικού αερίου από την ε, Ρωσία. Δεν σχολιάζω όμως την απόφαση αυτή. Αυτό που χρειάζεται η Βουλγαρία είναι ένας να απαλλαγεί από τη ρωσική κυριαρχία. Γι' αυτό και θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Σλοβακίας και να ξαναθέσει σε λειτουργία του σταθμού 3 και 4 του πυρηνικού της εργοστασίου. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειώσει τις ζημιές που ε, ε, παθαίνει από την κρίση αυτή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Α, μόλις τώρα ξεκίνησε το 2009. Επιτρέψτε μου να σας πω, λοιπόν, ότι δεν είναι συνηθισμένη χρονιά. Το 2009 θα γιορτάσουμε τα 20 χρόνια από το τέλος του ψυχρού πολέμου, από την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου και την λήξη του χωρισμού της Ευρώπης σε δύο μέρη. Σαν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και σαν Ρουμάνα που έχω ζήσει υποδικτατορία πρέπει να πω ότι για μας οι δύο δεκαετίες σήμαναν μετάβαση προς τη δημοκρατία και από τους άλλους αποδοχή των νεοφερμένων. Το 2009 θα πρέπει να είναι μια χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να πολεμήσουμε ώστε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη μοναδική για όλου του Ευρωπαίου πολίτε, ενιαία όπου και τα 500 εκατομμύρια άνθρωποι θα καταλάβουν ότι καλύπτονται τα δικαιώματά τους, είναι εγγυημένα, η αλληλεγγύη είναι πραγματική, δεν υπάρχει διάκριση κατά κανενός και κανείς δεν θα πρέπει να αισθάνεται ξένο σε μια Ενωμένη Ευρώπη. Είμαστε όλοι Ευρωπαίοι πολίτες, έχουμε τα ίδια συναισθήματα και τις ίδιες αξίες, ανεξάρτητα από που είμαστε το 1989. Το τώρα. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένος έχει συζητήσει οικολογικά θέματα. Να σας επιστήσω την προσοχή επί ενός θέματος που ενδιαφέρει τους νέους περιβαλλοντολόγους, οι οποίοι ήρθαν και μου το έθεσαν. Οι τιμές για το χαρτί και για το πλαστικό προς ανακύκλωση μειώνονται. Στην πολωνική αγορά επικρατεί τέτοια κατάσταση, ούτω ώστε εκείνοι που αγοράζουν χαρτί για ανακύκλωση λένε ότι είναι πολύ φθηνό. Εκείνοι που παράγουν το χαρτί, χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο χαρτί, λένε ότι αυτό το χαρτί είναι πολύ ακριβό. Άρα κάτι πρέπει να γίνει προ όφελο του περιβάλλοντο για να επιληθεί το πρόβλημα. Για την ώρα τα παιδιά μαζεύουν ανακυκλώσιμο χαρτί για εκπαιδευτικού λόγου, αλλά τελικά καταλήγει σε χωματερέ. Έκανα τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να πάρουν το λόγο στο δυνατόν περισσότεροι Τώρα σταματούμε εδώ τις παρεμβάσεις ενός λεπτού και ερχόμαστε στην ε, ε, μερίσια μας διάταξη η οποία προβλέπει την κοινή συζήτηση της έκθεσης της κυρίας Κρίστα Κλάς σχετικά με την οδηγία πλαίσιο για την ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων και την έκθεση της κυρίας Μπρέγερ σχετικά με την διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά οι συγγήτρες θα ξεκινήσουν τη συζήτηση. Πρώτη θα πάρει το λόγο η κυρία Κλάς για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Βασιλείου, κύριε Δήμα, εσείς κυρίες και κύριοι, σήμερα